chers Αγαπητοί συνάδελφοι, ας δούμε την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμά μας έτσι ώστε τα μέλη που το επιθυμούν, δηλαδή πλειοψηφία ελπίζω, να συμμετάσχετε στην κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Ελευθεριών Πολιτικών Ελευθεριών για την κατάσταση της Ευρώπης. Ο κύριος Ορί, από όσο γνωρίζω, θέλει το λόγο και, το δίνω, και τον δίνω. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. szeretnék egy kicsit többet hallani, hogy hogy is történt ez a, ez a módosítás. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στους συντονιστές την προηγούμενη εβδομάδα δεν μιλήσαμε για αυτό το θέμα. Βεβαίως κατανοώ τους λόγους, αλλά η, από όσο γνωρίζω υπάρχουν παράλληλες δραστηριότητες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν οι βουλευτές να συμμετάσχουν σε μια συνεδρίαση με τους συντονιστές και τους αντιπρόεδρους. Κανένας δεν ήρθε σε επαφή μαζί μου επί του θέματος. Με συγχωρείτε, αλλά δεν άκουσα την αρχή της παρέμβασής σας και δεν ξέρω πού αναφέρεστε. Μιλάτε για την τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης. Αυτό σας απασχολεί. Ναι, πρόκειται για την αλλαγή που έγινε επί της ημερήσιας διάταξης. Δεν θα ξεκινήσουμε μία συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τόμας Μαν, γιατί θα μας μιλήσει για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Μετά όμως θα συνεχίσουμε τις εργασίες όπως προβλέπονται. Δύναμη του κανονισμού. Η πρόεδρος ή ο πρόεδρος αποφαίνεται για τις δραστηριότητες και ενημερωθήκατε μόλις ελήφθη η απόφαση δεν ορίζουμε την ε, ημερήσια διάταξη στους συντονιστές. Κύριε Ορή, δεν ε, ε, ισχύει κάτι τέτοιο. Γνωρίζετε τη διαδικασία και ξέρετε ότι ποτέ δεν διαβουλευτήκαμε για την ημερήσια διάταξη για τις εργασίες. Η ευθύνη εναπόκειται στη γραμματεία μαζί με τους εισηγητές και τα μέλη που πρέπει να παρέμβουν σε σχέση με το θέμα που εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη. Θα δώσω το λόγο στον αντιπρόεδρό μας και μετά θα κλείσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Τόμας Μάν. Κυρία Πρόεδρε, ήθελα να πω κάτι για την ημερήσια διάταξη. Στηρίζω και εγώ αυτό που λέει ο κύριος Όρη. Η αλλαγή που έχει γίνει τώρα από τις 3 στις 4 ε, κάποιοι ε, ευρωβουλευτές θα εκπλαγούν. Κάποιοι που θα έρχονταν για να ε, παρακολουθήσουν το τι γίνεται με τις γνωμοδοτήσεις δεν θα το έχουν μάθει και εκτός αυτού, επειδή αφορά και εμένα, στην ημερήσια διάδοξη όπως, το, όπως την είχαμε, στις, 15, και στις 3 και 4 μέχρι τις 4 θα βλέπαμε τη δική μου έκθεση. Ε, και τώρα είναι, έχουμε, έχουμε, έχει μειωθεί ο χρόνος που είχα κατά 25 λεπτά και του κυρίου Κάσα επίσης. Οπότε έχουμε και λιγότερο χρόνο για να συζητήσουμε. Μας εκπλήσετε και με τις αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Ξεκινούμε και διαφορετική ώρα και δεν το έχουμε συζητήσει με κανέναν. Είναι κάποιοι που είναι έξω και θα έρθουν στις 3 κανονικά και στις 3 θα έχει τελειώσει η συνεδρίαση θα έχουν να συζητηθεί τα σημαντικά. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να περάσει έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Εντάξει, είναι σημαντικό να, να, να συζητήσουμε και την κατάσταση των Ρωμά, προφανώς, στην ε, ε, Ολομέλεια. Και γνωρίζουμε πραγματικά πώς έχει η κατάσταση. Φυσικά είναι λοιπόν θέμα αυτό προς συζήτηση, αλλά ε, απ' την άλλη να αλλάζουμε την ημερήσια διάταξη, να ξεκινούμε πιο νωρί. Να είναι, είναι πολύ ασυνήθιστο και πραγματικά και εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει ο κύριος Ορή. Κύριε Αντιπρόεδρε, είναι γεγονός ότι η κατάσταση αυτή είναι ασυνήθιστη αλλά η κατάσταση που γνωρίζουμε στην Ευρώπη είναι μια κατάσταση άκρος έκτακτη και έκριθμη και θα πρέπει να αποφανθούμε για την κατάσταση των Ρωμά. Γι' αυτό θα πρέπει να δείξουμε μια ευελιξία. Αυτό ακριβώς κάναμε και σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας γιατί θεωρώ ότι το γεγονός ε, ότι θα συμμετέχουν τέσσερις επίτροποι σε αυτήν την ακρόαση είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Αυτό το στοιχείο παρενέβη μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών και τη στιγμή που έπρεπε να γίνει μια διατησία, εσείς ενημερωθήκατε. Ε, από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τελειώσαμε με αυτό το σημείο λοιπόν. Θα ήθελα να σας πω ότι με βάση τον κώδικα δεοντολογίας... Όχι, το θέμα έχει λήξει. Η ομάδα σας αποφάνθηκε, είπατε, μιλήσατε για την ανησυχία σας. Δεν θα αλλάξουμε τη διαδικασία μέχρι τις 3. Αν θέλετε να επανέλθετε, θα επανέλθουμε κατά την προσεχή συνεδρίαση των συντονιστών. Κύριε Ορή, δεν θα ήθελα να λάβετε το λόγο, πραγματικά. μέσα στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας, της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας, ο κύριος Σέρκας μπορεί να μας πει πώς έχουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την πρόταση οδηγίας. Ο κύριος Σέρκας θα μας μιλήσει αύριο μετά την ψηφοφορία. Άρα εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Και φτάνουμε στις ανακοιώσεις της Πρόεδρου. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω την παρουσία της κυρίας Σίλντιγκο Καλπέλτς, ε, αναπληρώτηρας του ΕΛΚ, που ε, αντικαθιστά την κυρία Ενίκο Ζωρή. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κατά την παράδοση η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο και θα βρείτε και στο φάκελό σας την ανακοίνωση της Γραμματείας της Επιτροπής Απασχόλησης ως προς την διαδικασία προϋπολογισμού 2011 για τους οργανισμούς που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ε, της δικής μας ευθύνης. Η ανακοίνωση διατίθεται στα αγγλικά. Επίσης, στο φάκελό σας θα βρείτε την ανακοίνωση της γραμματείας. Πρόκειται για έναν κατάλογο που έχει καταρτήσει η γραμματεία, όπως ζήτησαν ορισμένε ομάδες, έτσι ώστε να δούμε ποιοι είναι οι ορισμοί που χρησιμοποιούμε ως Επιτροπή. Αυτή η ανακοίνωση διατίθεται στα αγγλικά. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι η ομάδα εργασίας για τα κοινωνικά ζητήματα που συνήλθε στις 24 Σεπτεμβρίου διαβίβασε στις μόνιμες αντιπροσωπείες τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση με τις τροποποιήσεις, τις τροπολογίες υπό την ευθύνη του κυρίου Τσαμπαωρή που αποτελούν στοιχεία κατά προτεραιότητα. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό στοιχείο μέσα στα πλαίσια της ε, έγκρισης των κατευθυντηρίων γραμμών από το Συμβούλιο και ελπίζω ε, αυτή τη στάση να ακολουθήσει και η Κόρεπερ και το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ. Κύριε Ορή, θέλετε να παρέμβετε ως εισηγητής, έχετε το λόγο. Όχι, δεν πρόκειται για αυτό το ζήτημα. επί του σημείου 4 Διακόπτη πρόεδρο. Έχω διαδικαστικό επί διαφορετικού θέματος. Πρέπει να δεχτείτε. Τη στιγμή που υπάρχει περισσότερο από ένα διαδικαστικό, κολλησιεργούμε και δεν μπορώ να το δεχτώ, εντάξει. Σημείο 4. Δημογραφική διακόπτη ο κύριος Όρη. Ο κύριος Τόμας Μαν έχει το λόγο για το σημείο 4 και με βάση τις 24 τροπολογίες συμβασμού για να προετοιμάσουμε την ψηφοφορία. Έχετε το λόγο για την οικονομική διακυβέρνηση. Ε, κυρία Πρόεδρε, είναι λίγο δύσκολο υπό τέτοιες συνθήκες να σας μιλήσω. Όταν ο συντονιστής δεν μπορεί να λάβει το λόγο μιας πολιτικής ομάδας, ε, σας είπα ότι είναι πολύ δύσκολο ε, αντί για 45 λεπτά να έχουμε 25 λεπτά στη διάθεσή μας για να συζητήσουμε το ζήτημα. Ε, αν δεν γίνει ε, προφορικά σήμερα, αν δεν προλάβουμε, θα πρέπει να δούμε τα σχόλιά σας γραπτός. Λοιπόν, για την έκθεσή μου υπήρξαν 253 ε, τροπολογίες. Ε, ε, τις τροπολογίες από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τι δέχομαι, τις οικονομικής, των οικονομικών υποθέσεων δεν μπορώ να τι δεχτώ, τι εξέτασα. τώρα, για, τους, για τις έχουν υπάρξει 20. Ε, που, με τις οποίες συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες, οπότε οι συνάδελφοι που ήταν ε, διατεθειμένοι να, τους, ε, να τις δεχθούν, παρακαλώ να τις δεχτούν. έλαβα πάρα πολλά τηλεφωνικά, τηλεφωνικές κλήσεις, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. για κάποιες τροπολογίες καταφέραμε να τις κάνουμε λίγο πιο μικρές. Επίσης, Υπήρξαν 74 τροπολογίε, οι οποίες επίσης είναι, μπήκαν στο κείμενο, ε, κάποιες αποσύρθηκαν. Τώρα, για την Άλντε είχαμε 50 τροπολογίε 43 έγιναν δεκτές. Μιλούμε για, την, ε, για, τις, ε, για μια νέα νομική βάση για να εξαλείψουμε την διακριτική μεταχείριση έναντι των ηλικιωμένων. Φυσικά πρέπει να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί άμεσα η οδηγία. Ε, συμφώνησα με πάρα πολλές ε, προτάσεις σας ε, και επίσης κάποιοι από τους ε, συντάκτες των, των, κάποιοι από τους συντάκτες συμφώνησαν μαζί μου. Επίσης από τους πρόεδρους είχα 48, τις 39 τις δέχτηκα. Προσπάθησα λοιπόν να καταλήξουμε σε, έναν ευρύ, σε μια ευρεία συμφωνία. Τα καταφέραμε πολύ. Καταφέραμε επίση να διαγράψουμε 133 α, τροπολογίες. Ξέρω ότι πρέπει να υπάρξουν κίνητρα για τους εργο, εργαζόμενους που είναι πάνω από, 60 ετών. Ε, πρέπει να έχουν και αυτοί τις δυνατότητες που πρέπει. να, είναι, να έχουν ε, σε πάση περιπτώσει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Δεν φτάνει. θέλουν να παραμείνουν στην, να λένε θέλω να παραμείνω στη δουλειά μου, αλλά πρέπει να τους δίνεται και η ευκαιρία να το κάνουν αυτό. Οπότε πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει ευελιξία. Και δεύτερον, Υπήρξε άλλο ένα θέμα για το όριο ηλικία για τη συνταξιοδότηση σε κάθε τομέα. Νομίζω ότι ε, παρά είναι αυτό. Ε, ίσως αυτό θα πρέπει να το αφήσουμε στους κοινωνικούς εταίρους, να δούνε δηλαδή ποιες είναι οι σωστές ρυθμίσεις, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχουν διαφορετικά όρια συνταξιοδότηση σε κάθε κράτος μέλος. το, είδαμε, το συζητήσαμε και στο Στρασβούργο αυτό αλλά και σε άλλε χώρε υπάρχουν διαφορετικά ε, όρια συνταξιοδότηση. Οπότε νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μπούμε σε τέτοια χωράφια. Για την ε, κυρία Πλάμπα από τους ε, σοσιαλιστές. Το βασικότερο πρόβλημά μου ήταν με την 126 και με την 129 τροπολογίες που υπέβαλε για την κατάργηση της πρόορης σύνταξης, της πρόορης συνταξιοδότησης η δική μου εμπειρία από τη δική μου χώρα όταν έγινε αυτή η, ε, όταν υπήρξε, εφαρμόστηκε αυτή η ε, συμφωνία, κάποιοι ναι, ε, συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα. Αλλά σε κάποια μέρη αυτό δεν εφαρμόστηκε. νομίζω ότι δεν θα πρέπει να, υποστηρίξουμε μια τέτοια διάταξη που να, υπο, να εισαγάγει την πρόωρη συνταξιοδότηση θα πρέπει να δώσουμε οικονομικά κίνητρα. Εγώ ε, είμαι υπέρ επιδοτούμενων προγραμμάτων ε, κρατικών. Τώρα για την κυρία Ράπτη. Θέμα των ε, εγγυήσεων για, τις, για τους έξι μήνες. Το συζητήσαμε από κοινού, το κάναμε τέσσερις, τέσσερις μήνες, δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν. Θεωρώ ότι όντως είναι σημαντικό το μήνυμα που έχουμε να δώσουμε ότι μετά από, τα τέσσερα, ε, μετά από τους τέσσερις μήνες ε, ανεργίας να δίνουμε στους ε, νέους την δυνατότητα να βρίσκουν θέση εργασίας ή να βρίσκουν θέση για περαιτέρω εκπαίδευση. Να τους δώσουμε λοιπόν ευκαιρίες και βεβαίως αυτό θα πρέπει να το κάνουν όλες οι επιχειρήσεις με τον ίδιο τρόπο και να υπάρχει δηλαδή και υποστήριξη και από τη μηχανία αλλά και από το κράτος. Από την ΚΟΕ τώρα 44 τροπολογίες, κάποιες τις ε, δέχομαι, της κυρίας Τσίμερ επίσης όλες τις δέχτηκα και του ε, συναδέλφου Λοχιαρικ. προβλήματα είχα με την συνάδελφο Higgins. Ζητά πολλά τα οποία δεν μπορώ να τα δεχτώ, δεν μπορώ να τα υποστηρίξω. Ας πούμε δημογραφική ε, μετανάστευση και συνέπειές της ε, ότι η οικογένεια είναι το πυρήνα της κοινωνίας. Εντάξει, δεν διαφωνούμε. Ε, προφανώς η οικογένεια είναι μια, μια, ο πυρήνας της κοινωνίας και πρέπει να τη χάνει και τις ανάλογες ε, μεταχείρισης. Τώρα, εκεί που λέει ότι πρέπει να διαγραφεί ο συμψηφισμός του προπολογισμού, δεν μπορώ να συμφωνήσω. Ε, εγώ θέλω να έχουμε ε, ευελιξία στην ε, πρότασή μας για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις πραγματικές ανάγκες. Τώρα, για τους πρασίνους, τις περισσότερες τροπολογίε τις δέχτηκα. Είχα 22 και δέχτηκα τις 20. 18 συμβιβαστικές. Ένα πρόβλημα μόνο είχα με την συνάδελφο Κορνέλισεν. Εγώ ανέφερα ότι θα πρέπει να έχουμε ε, μια ευρωπαϊκή εγγύηση για τους νέους, αλλά βεβαίως θα πρέπει να γίνονται από την άλλη πλευρά και προσπάθειες από τους ίδιους τους νέους. Προφανώς δεν γίνεται να πέφτουν σαν μάνα εξ τα προγράμματα για τους νέους. Προφανώς πρέπει και οι ίδιοι να κάνουν κάτι, πρέπει και οι ίδιοι να θέλουν να προσφέρουν και βεβαίως να τους δίνεται η αντίστοιχη ευκαιρία. Ε, νομίζω λοιπόν ότι ε, αυτό δεν μπορεί να λυθεί έτσι καλά μέσω ενός ε, συμβιβασμού. Επίσης, για τον ελάχιστο μισθό, για το ελάχιστο εισόδημα είχαμε μια διαφορά και έχω ζητήσει μια χωριστή ψηφοφορία, ψηφοφορία σε τμήματα για την 204. Ε, επίσης είχα δύο ε, τροπολογίες οι οποίες έγιναν κομμάτι συμβιβαστικών λύσεων Είπατε όμως ότι έχουν αυξηθεί τα όρια ε, των, της κληρονομιάς. Ε, πολλές φορές όμως ε, μιλούμε για θέσεις εργασίας που είναι ή χρονικά περιορισμένες ή πολύ ευαίσθητες. Ε, επίσης η φροντίδα των μικρών παιδιών όταν οι γονείς δουλεύουν είναι πολύ σημαντική. Συμπέρασμα. 22 συμβαστικέ προτάσεις. Πάνω από 80% των τροπολογιών έγιναν δεκτέ σε, πολλούς, σε πολλά τμήματα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό και σας ευχαριστώ όλους για την α, συνεργασία. Ήταν πολύ καλά η δουλειά που κάναμε. Θα σταματήσω εδώ γιατί χρόνο δεν έχουμε όπως είπαμε. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, euh, le Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κυρία ε, Κάστεξ καταρχήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαν για το πνεύμα συνεργασίας που τον διακατήχε για αυτή την έκθεση και για να φτάσουμε σε τροπολογίες συμβιβασμού. Νομίζω ότι προχωρήσαμε σε πολλούς τομείς συνενετικά και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Για να ολοκληρώσουμε τη συνεργασία μας υπάρχουν δύο προφορικές τροπολογίες στου συμβασμούς που μας απασχολούν και τους δύο. Πρόκειται για τον συμβασμό L για την διαβίου μάθηση, διαβίου κατάρτιση. Θα ήθελα να, να αντικαταστήσουμε το only με το specially σε σχέση με την κατάρτιση. Εάν συμφωνεί θα του διαβιβάσω σε αυτή την προφορική τροπολογία, η δεύτερη προφορική που του προτείνω αφορά το N, όπου μιλάμε ε, για το full employment, για population aged over 50. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ε, διατυπώσουμε κάπως διαφορετικά, δηλαδή να μιλάμε για αποζημίωση της τάξης του 55%. Έτσι ώστε να ορίσουμε, να διαφοροποιήσουμε την πλήρη απασχόληση με την μερική απασχόληση της τάξης του 55%. Θα ήθελα λοιπόν να αντικαταστήσουμε με το, το aiming δηλαδή που έχει ως στόχο μιλώντας για ένα ελάχιστο 55%. 55% απασχόλησης. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε με αυτή την προφορική τροπολογία. Θα σας την διαβάσω γραπτός. Όσον αφορά τις άλλες συμβιβαστικές τροπολογίες, Η σοσιαλιστική ομάδα δεν ε, ε, μπορεί να πει ότι συμφωνεί απόλυτα. Τις περισσότερες θα τις υπερψηφίσουμε. Όμως υπάρχουν αποκλήσεις μερικές. Και η απόκληση αυτή δεν ε, μειώθηκε σε σχέση με την ηλικία συνταξιοδότησης και της ε, ηλικία πέρα από τη συνταξιοδότηση, δηλαδή κατά πόσο μπορεί κανείς να αποσχολείται μετά από την ηλικία της νόμιμης συνταξιοδότησης. Ως προς το συμβιβασμό, την ε, τροπολογία συμβιβασμού μάλλον ε, J, θα την υπερψηφίσουμε εάν γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία το ξέρω ότι δεν γίνεται ξεχωριστή ψηφοφορία στις ε, τροπολογίε συμβιβασμού, αλλά τη στιγμή που δεν έχουμε προσυπογράψει αυτή την τροπολογία θα πρέπει, αν γίνει ξεχωριστή, να μπορέ, θα μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε ένα τμήμα, αλλιώ όχι. γιατί φαίνεται κάπως αντιφατική, δηλαδή το δεύτερο σκέλος ε, είναι αντιφατικό σε σχέση με το πρώτο. Διαφορετικά θα υπερψηφίσουμε την έκθεση, αν και σε ορισμένα ε, σημεία θα υπάρξει διαφοροποίηση. Η κυρία Λίν και μετά η κυρία Μπάουερ. Λίν. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον Τόμας Μαν για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο Σκιώδης για την ομάδα Άλντε. Ξέρω ότι χρειάστηκε να καταβάλεις ε, τεράστιες προσπάθειες και να εξετάσεις όλες αυτές τις τροπολογίες όπως έκανα και εγώ. Τιτάνιο το έργο και πιστεύω ότι πραγματικά τα κατάφερες πολύ καλά και έχεις ε, καταφέρει να καταλήξεις σε πολύ καλές συμβαστικές τροπολογίες. Έχω βέβαια δύο τρία σημεία στα οποία δεν διαφωνώ, ιδίω όσον αφορά το ζήτημα τη διακριτική μεταχείριση. Η τροπολογία 69. η οποία πέρασε και στην Ολομέλεια και η σχετική οδηγία για την ε, κατάργηση της διακριτικής μεταχείρισης προφανώς είχε ιδιαίτερη υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το μόνο το οποίο λέω είναι ότι θα πρέπει να διέπει η οδηγία αυτή και το πνεύμα αυτής εδώ της πρότασης. όσον αφορά τη συμβαστική όμικρον. Προτείνω να την καταψηφίσουμε γιατί προτιμώ το αρχικό κείμενο, την αρχική παράγραφο 13 δηλαδή. Θα κάνω μια σύσταση λοιπόν καταψήφισης της τροπολογίας αυτής γιατί θεωρώ όπως είπα ότι η αρχική διατύπωση ήταν πολύ καλύτερη. Συμβαστική τροπολογία 1. Δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη ούτε με αυτή Ωστόσο, πιστεύω ότι εφόσον συμφωνούν και οι υπόλοιποι, θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε επιπλέον τη δική μου τροπολογία 20. Δεν ξέρω αν η γραμματεία ή οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να δουν αν η 120 μπορεί να συνδυαστεί με την συμβαστική τροπολογία 1. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ένα τμήμα τουλάχιστον της 120 να περάσει στη συμβαστική τροπολογία 1. Το επιχείρημά μου είναι ότι καθότι δική μου τροπολογία δεν πέρασε στη συμβαστική N, θα μπορούσε τουλάχιστον επιπλέον να ψηφίσουμε με τροπολογία 120. Τώρα όσον αφορά την συμβαστική B, Β. Προτείνω να την καταψηφίσουμε έχει να κάνει με το ποιος ανατρέφει τα παιδιά. Νομίζω ότι αυτό δεν αποτελεί δική μα αρμοδιότητα ούτως ή άλλως. Το βασικό πνεύμα της τροπολογία δεν με βρίσκει αντίθετη, αλλά νομίζω ότι δεν είναι δική μα αρμοδιότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο βρίσκεται στο πλαίσιο αυτό. Η τι επίση νομίζω ότι υπερβαίνει τη δική μα αρμοδιότητα, γι' αυτό προτείνω να την καταψηφίσουμε. 175 τώρα. Δεν ξέρω αν ο συντάκτη τροπολογίας αυτή είναι παρόν, Κορνίλσεν. Είναι εδώ, η συνάδελφος. Ή να με εξηγήσει κάποιο τι θέλει να πει, κυρία Κορνέλσεν. αντικαθιστά μάλλον εισάγει τον όρο reconciliation, συμφιλίωση. Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε καν στα αγγλικά τι σημαίνει ο όρος αυτό στο, στα συμφραζόμενα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι θέλουμε, τι εννοούμε χρησιμοποιώντας τον όρο reconciliation στην ε, τροπολογία αυτή. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος συνάδελφος να με διαφωτίσει. Καταλαβαίνω πάλι ποιο είναι το βασικό πνεύμα πίσω από αυτή την τροπολογία, ότι δεν θέλουμε μόνο την οικογένεια, αλλά κάθε μορφή οικογενειακή σχέση μπορεί να υφίσταται. Θεωρώ πάντω ότι ο όρο reconciliation δεν σημαίνει κάτι, τουλάχιστον στα αγγλικά δεν σημαίνει κάτι στο πλαίσιο αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ και σε ευχαριστώ, Τόμα, πάλι για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Η κυρία Μπάουερ, καταρχήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που άφησε το θέμα η κυρία Λίν. Ε, προετοίμασα την γνωμοδότηση από την Επιτροπή ΦΑΜ. Η συμφιλίωση της οικογενειακής ζωής με την επαγγελματική είναι ένα θέμα κλειδί. Η απασχόληση των γυναικών μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. 20 όρισε στόχους που είναι αδύνατοι αν δεν λάβουμε υπόψη τους διαφορετικούς οργανισμούς και τα διάφορα κοινωνικά στρώματα. Χρειάζονται πολλά μέτρα από επίπεδο εργοδοτών μέχρι τις τοπικές αρχές, τις περιφερειακές αρχές. Θα πρέπει να ληφθεί πληθώρα μέτρων, διότι πολλές φορές υπάρχει επικάλυψη οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Υπάρχει μία σειρά ε, υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτούς τους τομείς και αφορούν ιδιαίτερα τις γυναίκες. Εάν δεν μπορούμε να μειώσουμε αυτές τις υποχρεώσεις ε, δημιουργώντας ένα καλό υπόβαθρο θα είναι αδύνατον να αυξηθεί η γυναική απασχόληση όπως έχει οριστεί από την στρατηγική 2020. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τόμας Μαν για αυτή την εξαιρετική εργασία. Είναι γεγονός ότι οι τροπολογίες που συντάξαμε στη γνωμοδότηση δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να λάβετε όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τόμας Μαν για την κατανόησή του. Η κυρία Μωρέ. Θα συνεχίσω το σκεπτικό της κυρίας Μπάουερ με βάση ορισμένες τροπολογίες οι οποίες ε, υποβλήθηκαν ως συμπλήρωμα του κειμένου του Τόμας Μαν το οποίο είναι ένα πλήρες κείμενο. Πέρα από το κείμενο αυτό Οι τροπολογίες αναφέρονται στο γεγονός ότι για να συμφιλιώσει κανείς την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή, για να υπάρχει δηλαδή η ισότητα των πολιτών στην Ευρώπη, ε, προτάθηκαν τροπολογίες που ζητούν να μην υπάρχει μισθολογικός περιορισμός σε σχέση με την μείωση του ωραρίου που σχετίζεται με τις οικογενειακές επιβαρύνσεις. Νομίζω ότι σωρευτικά μερικές τροπολογίες διαστρεβλώνουν το στόχο μας, διότι πίσω από την απασχόληση των γυναικών τι θέλουμε, θέλουμε ισότητα στις σταδιοδρομίες. Βεβαίως μας ενδιαφέρει και η μισθολογική ισότητα, αλλά αυτό το οποίο είναι πολύ σοβαρό και το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι μετά τη γέννα, τη μητρότητα, τα οικογενειακά βάρη δεν υπάρχει ισότητα στη σταδιοδρομία. Γι' αυτό προσδίδω μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα και θα ήθελα ο Τόμας Μαν να ενσωματώσει αυτή την ιδέα σε μία από τις τροπολογίες του. Δηλαδή θα μπορούσε να ενταχθεί στην 178 για τους άντρες και τις γυναίκες της κυρίας Όμεν Ρόιτεν ή σε άλλες ε, τροπολογίες, σε κάποια άλλη τροπολογία ενδεχομένως. Την 185, στην παράγραφο 25. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να ορίσουμε το θέμα της ισότητας στην σταδιοδρομία σε αυτή τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τόμας Μαν για την υπέροχη εργασία του επί ενός θέματος που μας απασχολεί όλους. Και ελπίζω αυτό το θέμα, να, αυτή η έννοια να ενσωματωθεί στις σκέψεις μας. Τσάπνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω Τόμας για την πολύ σημαντική εργασία. Το θέμα της γύρανσης του πληθυσμού θα μας απασχολεί πολύ χρόνο, για πολύ χρόνο. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η γύρανση του πληθυσμού αλλάζει τον κόσμο, όπως το ζούμε. Χαίρομαι διότι ο Τόμας μας έδωσε τη δυνατότητα να εξετάσουμε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να μας απασχολήσει η ισότητα δικαιωμάτων σε όλη την κοινωνία και στα διάφορα συστήματα. Οι πολιτικοί θύνοντες θα πρέπει να αντιδράσουν σε αυτή την πραγματικότητα. Δεν μπορούν όμως να μας ε, υποσχεθούν κάτι το οποίο δεν μπορεί να πληρωθεί. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κοινωνική ασφάλιση ε, η οποία θα είναι ικανοποιητική οικονομικά. Θα πρέπει να γίνει μια μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό και αυτό αφορά και τις κοινωνικές παροχές. Γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ηλικιωμένους στην, ε, σε αυτή τη φάση της ζωής τους θα πρέπει να συμφιλιώσουμε την οικογενική ζωή και να υπάρχει ε, και πλήρωση του χάσματος μεταξύ των γενεών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τόμας για τη συνεργασία. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Πριν όμως, θα ήθελα να σας ενημερώσω για την παρουσία δημοσιογράφων που πραγματοποιούν το WebDoc και θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή η δυνάμη του, της τροπολογίας 120 όπου η κυρία Ελίζα Μπεθλίν σας ζήτησε να δεχτείτε την τροπολογία ως προσθήκη στην πρόταση συμβασμού N να λάβουμε υπόψη το πρώτο μέρος της προσθήκης της πρότασης ΛΙΝ που είναι συμβατό, δηλαδή να ισχύσει ευρωπαϊκή νομοθεσία που να απαγορεύει τη διάκριση με βάση την ηλικία. Ε, θεωρήστε το ως προσθήκη και αφήστε το δεύτερο μέρος. Δηλαδή να μιλάμε για την ηλικία συνταξιοδότης που πολλές φορές ορίζεται αυθαίρετα, διότι έρχεται σε αντίθεση με τον, την πρώτη συμβασμό όπως την έχετε προτείνει. Δίνω το λόγο στον εισηγητή. Äh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ευχαριστώ και για την στήριξή σας. Νομίζω ότι από κοινού καταλήξαμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα γνωμοδότηση που είναι αρκετά καινούρια γιατί δεν βλέπει μόνο το θέμα της ηλικία ή μόνο το θέμα των νέων αλλά ε, έχει μια προσέγγιση και για τα δύο. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή και η συζήτηση στο Στρασβούργο και η ε, συζήτηση που κάναμε στις ομάδες. Ε, η συνάδελφος Κάστεξ. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Οι δύο προφορικές σας ε, ε, τροπολογίες, ε, Φρανσουάζ, εντάξει, αποδεκτές μπορούν να γίνουν και για την, αντί για only να πούμε specially, δεν είναι πρόβλημα αυτό, αλίμονο. Θα το δω βέβαια για να είναι καλή και η διατύπωση, αλλά έχω καταλάβει τι εννοείς και δεν υπάρχει πρόβλημα. για το 55% minimum που είπες να συμπεριλαμβάνουμε. θα πρέπει να το συμπληρώσουμε Όλοι θα θέλαμε να είναι πολύ μεγαλύτερη η απασχόληση και φυσικά δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι λιγότερο. Θα δω λοιπόν πώς μπορώ να το εντάξω μέσα στην, μέσα στην διατύπωση. Για, το, για την συμβαστική G, κατάλαβα τι θέλεις με την χωριστή ψηφοφορία. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα προφανώς. νομίζω όμως ότι μέσω των συμβασμών έχουμε πετύχει πολλά. Για την ε, ε, διακριτική μεταχείριση προφανώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα να έχουμε μία επιπλέον ρύθμιση, ε, ίσως καλό θα ήταν ε, να έχουμε να έχουμε εφαρμόσει και άλλε διατυπώσει που υπάρχουν, άλλε διατάξει που, έχουν, που, έχουν θέμα, που, που θέτουν θέμα ε, εφαρμογή. Όχι να εφευρίσκουμε απλώ καινούριε, να εφαρμόζουμε κάποια στιγμή και αυτέ που ήδη υπάρχουν. Την 13 ε, εντάξει μπορώ να την ε, υποστηρίξω. Ε, ε την, δεν μπορώ να τα δεχτώ όλα, καταλαβαίνετε. Συμβιβασμού κάνουμε, δίνετε κάτι εσεί, δίνω κάτι κι εγώ, για να καταλήξουμε σε μια λύση που να μας ικανοποιεί και τους δύο. Τώρα, ε, συμβαστική πρόταση νη. Να προσθέσω τα 120. Ε, θα το ξανασυζητήσουμε, θα έρθουμε σε επαφή και το απόγευμα, θα το, θα το δω. Και για, το, για τη συμβαστική 75, Βασικά η δική μας ε, άποψη είναι προφανώς να συνδυάζεται η επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. συμφωνώ με όλα όσα είπαν οι γυναίκες ε, και για τη συνάδελφο Μωρά ε, θα δω, θα δω τι μπορούμε να κάνουμε για την 178 και την 158. Θα, θα δω με ποια διατύπωση μπορώ να τα συνδυάσω ε, για να σας ικανοποιήσω. Ε, ευχαριστώ για την υποστήριξη λοιπόν. Και για τις κοινωνικές υπηρεσίες είναι σημαντικό αυτό που είπες γιατί όντως ε, χρειάζεται να αναφέρεται και αυτό. Η πρώτη τώρα της Προέδρου για το 120 να, να, το, να το παραλείψουμε από το κείμενο. Θα το κοιτάξω, αλλά θεωρώ ότι με όλες αυτές τις προτάσεις έχουμε μια πάρα πολύ καλή βάση για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιγητά. Μπορούμε λοιπόν αύριο να ψηφίσουμε, πιστεύω, χωρίς κανένα πρόβλημα. Αύριο λοιπόν κατά την πρωινή μας συνεδρία θα γίνει ψηφοφορία. Περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συντάκτη γνωμοδότηση, τον κύριο Ντέβιτ Γκάζα, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την αξιολόγηση που έκανε των 40 τροπολογιών, καθώς επίσης και των δύο συμβαστικών τροπολογιών που κατάφερε να συντάξει. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση την οποία θα ψηφίσουμε αύριο, αν όλα πάνε καλά. Είναι σημαντικό το ότι συζητάμε σήμερα τη γνωμοδότησή σας κύριε Κάζα γιατί σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει μια πολύ σημαντική πρόταση όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση και βλέπουμε επίσης ότι έχουμε και μια πολύ σημαντική πανευρωπαϊκή απεργία στις Βρυξέλλες η οποία συνδέεται και αυτή με την οικονομική διακυβέρνηση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. στις 4-5 Οκτωβρίου θα εγκριθεί στην ε, αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή η έκθεση, η έκθεση του κυρίου Φεϊό. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε και εμείς το χρόνο να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την έγκριση αυτής της γνωμοδότησης. Κύριε Κάζα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μ' άρεσε πολύ να λαμβάνω το λόγο παρουσία δημοσιογράφων Παρ' όλα αυτά δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να τροποποιηθεί η ημερήσια διάταξη. Πρότεινα εγώ μια αλλαγή και δεν μας δώστε τη δυνατότητα να εξηγήσουμε το διαδικαστικό αυτό αίτημα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι απαράδεκτο κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω να μην επαναληφθεί αυτό στο μέλλον. Γιατί δεν είναι σωστό ο Προεδρεύων σε μία επιτροπή να μην ακούει ένα αίτημα διαδικαστικό το οποίο μπορεί να έχει ένας συνάδελφος. Ναι, είπατε ότι είναι σημαντικό ότι συζητάτε σήμερα η έκθεση αυτή. Είχαμε πολλές τροπολογίες στη γνωμοδότηση αυτή και είμαι υπέρ των περισσότερων από αυτές. Οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί δίνουν μια προστιθέμενη αξία στην γνωμοδότησή μου και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σε θέση να τις δεχτώ. κυρία Γκρούνη Κοφεράτη στην παράγραφο 3 είχαν υποβάλει κάποιε τροπολογίε όσον αφορά την δημοσιονομική αξιολόγηση. Καταφέραμε να βρούμε μια συμβαστική λύση και είπαμε ότι θα πρέπει στην αξιολόγηση αυτή να λαμβάνουν υπόψη τα συνταξιδοτικά συστήματα. Πρέπει τα συστήματα αυτά να είναι όχι μόνο βιώσιμα, πρέπει να είναι τα κατάλληλα και τα πιο ασφαλή για του Ευρωπαίου πολίτες. Όσον αφορά την παράγραφο 7, που έχει να κάνει με το σύστημα κυρώσεων. Εδώ πέρα πάλι βρέθηκε μια συμβαστική λύση, ήταν πιο δύσκολο όμως αυτή τη φορά. Γίνανε διαπραγματεύσεις και καταλήξαμε στο ότι τα συστήματα κυρώσεων θα πρέπει να αποκλείουν τα διαρθρωτικά ταμεία και δεν θα πρέπει να προβλέπεται ένα περιορισμό εδώ πέρα στην ε, εκπαίδευση. Τα συστήματα κυρώσεων επίσης δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τα κράτη-μέλη από τη δημοκρατική συμμετοχή στη δικασία λήψη αποφάσεων. Χαίρομαι με την συμβαστική αυτή τροπολογία και ελπίζω το Κοινοβούλιο θα καταφέρει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα προ τα έξω. Επίση, έχουμε κάποιε τροπολογίε που έχουν να κάνουν με την ε, πρακτική αποδοχών στα πλαίσια του χρηματοπιστωτικού τομέα και ότι δεν θα πρέπει το σύστημα αποδοχών και μισθών να θέτει εν κινδύνο την ε, οικονομική διακυβέρνηση και τη σταθερότητα του συστήματο. Επίση, θέλουμε αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα. Έχουμε μία ξεχωριστή τροπολογία γι' αυτό. Στατιστικά δεδομένα που να αφορούν και την απασχόληση και να υποβάλλονται εγκαίρως. Αυτά είχα να σας πω, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Καλύτερα να σταματήσω στο σημείο αυτό και ευχαριστώ τους και ηγητές για την υποστήριξή τους, καθώς επίσης και όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής αυτής, οι οποίοι βοήθησαν στην, στο να καταλήξουμε συμβαστικές τροπολογίες. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κύριε εισηγητά. Έχουμε χρόνο, είχαμε χρόνο για να ακούσουμε τα επιχείρηματά σας και να ακούσουμε και την, απαντή, την απάντησή Κύριε Ράπτη, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά που έκανε, διότι αν δεν έχει κανείς ένα καλό κείμενο βάσης, δεν μπορεί να κάνει και τροπολογίες που να βοηθούν. Ε, ευχαριστώ επίσης τους άλλους συναδέλφους και όδους εισηγητές για την συνεργασία. Ε, αισθάνομαι ικανοποίηση για την συμβιβαστική δύο η οποία βάζει ζητήματα που εξυπηρετούν την κοινωνική διάσταση της οικονομικής διακυβέρνησης. Αισθάνομαι επίσης την ανάγκη να επισημάνω ε, ζητήματα τα οποία έχουμε επισημάνει και με την πρόεδρο της Επιτροπής μας, την κυρία Μπερές, σε κοινέ τροπολογίες που έχουμε καταθέσει και που αφορούν μεταξύ άλλων τη συμπερίληψη των στόχων της απασχόλησης, τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ εθνικών προγραμμάτων σύγκλησης, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τη στρατηγική της Ευρώπης 2020 και των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση, είναι πολύ σημαντικό επίσης το θέμα της ενεργοποίησης της οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας της συνθήκη της λισαβόνας ε, το θέμα των κυρώσεων ο τρόπος με τον οποίο ε, αντιμετωπίζεται στη συμβιβαστική ε, μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι θα μπορέσει η κοινωνική διάσταση των επιπτώσεων να είναι πραγματικά όσο το δυνατόν μικρότερη και βεβαίως να επισημάνω για μια ακόμη φορά το θέμα της ανάγκης υψηλής ποιότητας απασχόλησης. Τέλος κλείνοντας, ε, να καταθέσω και εγώ τη σκέψη μου για την διαδικασία και να πω ότι πραγματικά αισθάνομαι ότι σε κρίσιμες περιστάσεις όπως αυτές που ζούμε σήμερα, νομίζω ότι κάποιες φορές πρέπει να αφήνουμε την ουσία να έρχεται πρώτα, κύρια και πάνω από τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Euh, Ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Κύριο Έλμερ. Uh, Ευχαριστώ. Και πριν αναφερθώ στην έκθεση Κάζα, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τους συναδέλφους με, ως προς τα δρακόντια μέτρα ε, με τα οποία, όπως αντιμετωπίζετε δηλαδή τους βουλευτές και πώς προεδρεύετε. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ σε δύο-τρεις τροπολογίες. Στην τροπολογία 4 όπου λέμε ότι το κοινωνικό μοντέλο, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο αποτελεί ένα βασικό στοιχείο ανταγωνισμού. Θα ήθελα να είμαι σίγουρος ότι φοράω τα γυαλιά μου. Πιστεύουμε ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο αποτελεί προσόν για το διεθνή ανταγωνισμό. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό ε, μοντέλο αυξάνει το εργασιακό κόστος και το κόστος για την κοινωνική ασφάλιση. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε κατά πόσο ε, είναι σωστό να καταβληθεί το αντίτιμο αυτό. Αλλά το να πείτε ότι είναι προσόν το να αυξάνουμε το εργατικό κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δείχνει οικονομικό αναλφαβητισμό. Είναι το πιο τερατώδες πράγμα που έχω ποτέ διαβάσει στο Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό. Στη συνέχεια, ως προς την 22, όπου μιλάμε για μια ε, επιτροπή ψηλού επίπεδου. Όταν μιλήσουμε για την κοινωνική απάτη, βλέπουμε ότι μιλάμε για μία οργάνωση τύπου στάζη η οποία μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιβάλλει τις θέσεις της. Αυτή είναι μία πρόταση που μας σοκάρει. Πέρα από το ότι δημιουργούμε περισσότερες επιτροπές για εποπτεία των πάντων, αλλά η 25 είναι η πιο ανησυχητική γιατί μιλάμε για συντονισμό μισθολογικού. Το τελευταίο που θέλουμε, αν είμαστε ανταγωνιστικοί, είναι ο συντονισμός μισθών. Γιατί όλοι τι θα κάνουν, θα πάνε στις ε, χώρες χαμηλότερου εισοδήματο και θα επιβάλλουμε ε, κανόνες έτσι ώστε κανείς να μην εφημερεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν θα μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί την ε, χαμηλότερη μισθολογία. Λυπάμαι αν επαναλαμβάνω τα ίδια, αλλά αυτά που κάνουμε δεν είναι για την απασχόληση, αλλά για την ανεργία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ επιτυχή στο να δημιουργεί ανεργία και δυστυχώς δεν δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Κρότσμαν. Και μετά ο κύριο Ντερόζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, να συγχαρώ τον... Ε, και να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κάζα για τη δουλειά του έχει πραγματικά υποβάλει μια εξαιρετική ε, γνωμοδότηση, ταιριάζει, είναι σύμφωνη και η Επιτροπή Εκών γι' αυτό. Όντως ε, πρέπει να τηρήσουμε αυτά που συμφωνούνται, ώστε να έχουμε ε, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ή να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, νέα ανάπτυξη Τώρα, για τα οικονομικά δεδομένα των ε, εθνικών κρατών θα ήθελα να πω κάτι. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια, ε, περιβαλλοντικά κριτήρια που προτείνονται και σε κάποιες τροπολογίες. Υπάρχουν εξαιρέσεις για, την, μεσοπρόθεσμη, για τις μεσοπρόθεσμες συνέπειες. Τώρα, ένα υπερχρεωμένο κράτος ε, θα είναι σαφές δεν μπορεί να δώσει ούτε κοινωνικέ πρόνοιες γιατί δεν θα μπορεί κάποια στιγμή να τις καταβάλει. Οπότε είναι σημαντικό να ξεφύγουμε από όλες αυτές τις, από τις υπερχρεώσεις ώστε στο μέλλον να μην υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις κρατών που είναι υπερχρεωμένα. Γι' αυτό σήμερα ήδη πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι όλες αυτές οι, όλα αυτά τα χρέη που έχουν τα, τα κράτη ε, να μπορούν να αντισταθμιστούν παρόλα αυτά με, κοινωνικές, ε, με κοινωνική πρόνοια. Φυσικά πρέπει να φροντίσουμε την ε, κοινωνική συνοχή. Θα Πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο εάν δούμε αυτό το, σήμα, το σημείο με το συμψηφισμό που αναφέρεται. Τώρα, να δημιουργούμε συνέχεια νέες ομάδες ε, με εμπειρογνώμονες, με σοφούς κτλ. δεν νομίζω ότι θα λύσει το πρόβλημα. Ε, πρακτικές πρέπει να είναι οι λύσεις που θα επιλέξουμε. Για το λόγο λοιπόν αυτό λυπούμε που το, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τη συμβαστική πρόταση για την παράγραφο 7 γιατί νομίζω ότι περιλαμβάνει πάρα πολλές εξαιρέσεις. Ευχαριστώ όμως τον κύριο Κάζα που δέχτηκε και συζητήσαμε κάποιες από τις τροπολογίες και την ευελιξία που έδειξε για να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις. Εγώ δεν είμαι υπέρ, δεν είμαι υπέρ της, του συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως αναφέρεται στην έκθεση. η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να συμπεριλάβει και τις εθνικές ε, κυβερνήσεις. Ε, όλα τα υπόλοιπα δεν μπορούν να ισχύσουν. Συμφωνώ με αυτό που λέει η κυρία Χόκκιν ότι οι, κυρίσεις, κυρώσεις συγγνώμη, θα πρέπει να, να ειδωθούν και με το τι συνέπειες θα έχουν στους εργαζόμενους. Αυτά από μένα και ευχαριστώ. Ο Ντερόζα. Ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Ο κύριος Ντερόζα. Και μετά ο κύριος Κάζα για τα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό το ότι ζητάμε σήμερα την ε, γνωμοδότηση όταν κάνει τις έξι προτάσεις σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Οικονομική Διακυβέρνηση. Τέσσερις εκ των οποίων θα πρέπει να εγκριθούν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της συναπόφασης και θα πρέπει να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας για τις ε, υπόλοιπε. Είναι σημαντικό λοιπόν να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον από τη δική μα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ότι δεν είναι δυνατό να έχουμε μία αξιοπρεπή κοινωνία η οποία να βασίζεται απλώς στις έννοιες του ελλείμματος και η οποία να βασίζεται απλώς σε κάποια αυθαίρετα ή τεχνητά κριτήρια. Δεν μιλάω κατά της οικονομικής εξυγίανσης βέβαια. Αυτό το οποίο λέουν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο οικονομία. Ευρώπη σημαίνει και κοινωνία, ευρωπαϊκή κοινωνία. Επομένως τα επιχειρήματα που εξέθεσαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές δεν αντικατοπτρίζουν τους πραγματικούς λόγους οικονομικής κρίσης που διανύουμε. αναφερθήκαμε στην ε, γνώση οικονομικών στοιχείων από τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι όμως τελικά προωθούν όλο και περισσότερο την οικονομική απελευθέρωση, την κατάργηση των οικονομικών ρυθμίσεων. Θεωρώ ότι ακριβώς αυτά τα στοιχεία μας οδήγησαν στην οικονομική κρίση. Εξαιτία δηλαδή όλων αυτών των δαπανών που κάνανε οι τράπεζες και οι μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ετέθησαν κινδύνο και σε πάρα πολλές περιπτώσεις χάθηκαν ε, τα περιουσιακά στοιχεία των ίδιων των Ευρωπαίων πολιτών. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε εδώ πέρα μια ευρωπαϊκή οικονομία η οποία να λαμβάνει υπόψη της τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών. Δηλαδή αξιοπρεπείς κοινωνικές υπηρεσίες και ανάγκη για απασχόληση. Θεωρώ ότι οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προσπαθούν αυτή τη στιγμή ή δεν καταβάλουν ε, τι κατάλληλε προσπάθειε ή αρκετέ προσπάθειε για να πετύχουν τη λεπτή αυτή ισορροπία ανάμεσα σε οικονομία και κοινωνία, προστασία τη κοινωνία. Αναφερόμαστε εδώ πέρα, σε, αναφέρονται σε διάφορα ποσοστά, σε ένα 6%, σε συγκεκριμένου οικονομικού στόχου μείωση του ελλείμματο κάθε φορά, χωρί να λαμβάνουν υπόψη του άλλε κοινωνικέ πτυχέ, όπω για παράδειγμα η περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση, η φροντίδα των παιδιών κ.ο.κ. Θα ήθελα λοιπόν να στείλουμε το μήνυμα αυτό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τουλάχιστον το μήνυμα το οποίο στέλνουμε από την ομάδα των σοσιαλιστών είναι ότι η στάση τους δεν είναι ακόμα επαρκή και ότι θα πρέπει σαφώς να καταλήξουν σε μια συμβαστική πρόταση αν θέλουν να συναποφασίσουμε, αν θέλουν να συναποφασίσουν μαζί μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόεδρος, νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, άρα δίνω το λόγο στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως βλέπετε πολλές ε, τροπολογίες ε, έχουμε και έπρεπε και εγώ να καταλήξω σε κάποιες συμβαστικές. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν, ακόμα και από τον ίδιο τον Ρότζερ, ο οποίος αναφέρθηκε στην τροπολογία υπαριθμών 25 για τον συντονισμό της πολιτικής μισθών. Εγώ θα ήθελα αρνητικό πρόσημο στο σημείο αυτό, δεν συμφωνώ μαζί του. Όσον αφορά την τροπολογία 4 της κυρίας Μπέρες, European Social Model, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. Ο όρος αυτός είναι λίγο αμφίσιμος στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Το... Δεν είμαι κατά προφανώς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, αλλά νομίζω ότι δεν ταιριάζει πάρα πολύ καλά στο σημείο αυτό. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι μπορούμε να την υπερψηφίσουμε, όποιος βέβαια διαφωνεί θα την καταψηφίσει. Θεωρώ εν γέννη ότι η γνωμοδότηση αυτή όπως τροποποιήθηκε είναι μια καλή γνωμοδότηση θα Πρέπει βέβαια να έχουμε μια θετική έκβαση αύριο και πρέπει να σας πω ότι στι τελευταίε μέρε και ώρες κατάφερα να καταλήξω σε κάποιε θετικέ συμβαστικέ τροπολογίε. Πρόεδρο. Πολύ ωραία. Θα ψηφίσουμε αύριο τη γνωμοδότησή σας. Κύριε Σιγητέ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό τη μερίσια διάταξη. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 6 λέει πρόεδρο, όπου έχουμε εδώ πέρα του συντάκτε μιας μελέτης την οποία εμεί ζητήσαμε για το ρόλο της κοινωνικής προστασίας ως οικονομικού σταθεροποιητή. Άνω κάτω τελεία, διδάγματα της σημερινή κρίσης. Δεν ξέρω αν ο κύριος Έλμερ θα βρει μια απάντηση στο ερώτημα το οποίο έθεσε πριν από λίγο. Πάντως θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό το οποίο έθιξε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Βέρνερ Άισχολ, τον κύριο Ντόμας Λεωνί, τον Μάρτιν Ζεράρ και τον Μάτια Ντόλ, όλου του συντάκτε δηλαδή τη μελέτη αυτή που συνέβαλαν πολύ στι εργασίε τη Επιτροπή μα και να δώσω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Βέρνερ Άιχορστ για την παρουσίαση του πορίσματο τη μελέτη αυτή. Έχετε το λόγο. Okay, thank you very much. Uh, dear chairman, dear... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, Δυστυχώ ο κύριο Λεόνι δεν μπορούσε να έρθει σήμερα λόγω τη απεργία τη Βρυξέλλε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορέσουμε να σα παρουσιάσουμε την πρόσφατη μελέτη που κάναμε για το ρόλο τη κοινωνική προστασία ω οικονομικού σταθεροποιητή. την έρευνα αυτή την ε, ζήτησε η Επιτροπή σας και αναλύει αυτά που γνωρίζουμε για τον ρόλο του συστημάτων κοινωνικής προστασίας και των ιδιαίτερων διακριτικών μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο για την προστασία της αγοράς εργασίας και της οικονομίας του σύνολό της. Η έκθεση ξεκινά με μια περίληψη των υπαρχόντων ευρημάτων της κοινωνικής προστασίας ως οικονομικού σταθεροποιητή, βλέπει ποιες είναι οι συνθήκες κατά τις οποίες λειτουργούν ε, αυτά βλέπουν πώς, πώς μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικά τα μέτρα ώστε να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε και την α, οικονομία μέσω και οικονομικών αλλά και φορολογικών πολιτικών. Η έκθεση κάνει ένα διαχωρισμό μεταξύ των μέτρων διακριτικής ευχέρειας που έχουν τα κράτη-μέλη και των α, σταθεροποιητικών μέτρων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα κοινωνικά συστήματα, ε, ενώ τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας ε, εισάγονται λόγω της οικονομικής κρίσης ε, που βιώνουμε για να σταθεροποιήσουν την οικονομία. Είναι έκτακτα και τα ευρήματά μας δείχνουν ότι περίπου τα δύο τρίτα των μέτρων αυτών ε, αφορούν με θέματα κοινωνικής πολιτικής τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζω ότι αντέδρασαν άμεσα και συλλογικά ώστε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες αυτής της οικονομικής ύφεσης ε, και στην αγορά εργασίας και στην ε, πραγματική οικονομία. Αυτά για την ε, πολιτική αυτή που αφορά τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας θα δείτε ένα, μια συνολική καταγραφή των μέτρων αυτών που υπάρχουν που εγκρίθηκαν από το 2008 ε, μέχρι το 2010 με ιδιαίτερη αναφορά σε συγκεκριμένες πολιτικές, σε επιδόματα ενεργείας ε, σε, ενεργή, σε πολιτικές για την αγορά εργασίας, ώστε να, και με πολλά στοιχεία ώστε να είναι πιο κατανοητά τα πράγματα. Και βεβαίω τα σημαντικά μέτρα που έχουν ε, υιοθετηθεί σε ό,τι αφορά την ε, φορολογική μείωση, ώστε να σταθεροποιηθεί η αγορά εργασία. Μπορείτε λοιπόν να βρείτε μια γενική εικόνα όλων αυτών. Και εκτός αυτού θα δείτε και έναν υπολογισμό των, ε, των επιπτώσεων που είχαν, των συνεπειών που είχαν αυτά τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας στο ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη της και στην ε, απασχόληση. Είδαμε πολύ σημαντικές συνέπειες όταν ε, λάβαμε υπόψη και την διάδραση των μέτρων αυτών ε, και στα πακέτα φορολογικής ενίσχυσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία, υπάρχει λοιπόν συσχετισμός μεταξύ των ανοιχτών οικονομιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εσωτερική αγορά. Οπότε έτσι είναι πιο αποτελεσματικές οι πολιτικές. Από το να προσπαθούσαμε να τις εφαρμόσουμε σε μεμονωμένη βάση. Τα μέτρα αυτά διακριτική ευχαίρεια σταθεροποιούν τι θέσει εργασία, βοηθούν να δημιουργηθούν περαιτέρω θέσει εργασία κατά τη διάρκεια τη ύφεση και ένα ακόμη σημαντικό θέμα που αφορά τα μέτρα αυτά είναι το θέμα του χρονισμού. Δηλαδή πότε λαμβάνονται οι αποφάσει, πότε εφαρμόζονται οι αποφάσει που λαμβάνονται, ε, και αυτό είναι το κεφάλαιο που θα καλύψει εδώ ο συνάδελφος, ο Μάρκ. Ευχαριστώ. Για το χρονισμό των ε, μέτρων αυτών υπάρχουν κάποιες ε, σημαντικές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ειδικά η σωστή χρονική στιγμή των ενισχύσεων και η προσωρινή φύση τους. Δηλαδή δεν μπορούν να κρατήσουν, να διαρκέσουν για πάντα γιατί αλλιώς δεν θα αντιστάθμιζαν την κρίση θα την ενίσχυαν. Οπότε δεν θα ενίσχυαν την, ε, την έξοδο από την ύφεση. Υπάρχουν κάποια θέματα με το χρονισμό, τα, γιατί τα μέτρα αυτά θεωρούνται προβληματικά, επειδή υπάρχει ακριβώς αυτό το θέμα του χρονισμού. Δηλαδή τα κενά που υπάρχουν όταν η πολιτική ε, εφαρμόζεται Υπάρχει η εξωτερική πτυχή η οποία ε, μελετά τα δεδομένα, τα αποτελέσματα, συγγνώμη, αλλά υπάρχει και η εσωτερική πτυχή η οποία μελετά την εσωτερική διαδικασία. Και αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. Γι' αυτό αυτά τα μέτρα διακριτική ευχέρεια ε, θεωρούνται λιγότερο επιτυχημένα από άλλα σταθεροποιητικά μέτρα. Like Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η οικονομική ενίσχυση για τα διάφορα κράτη-μέλη. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά θετικά για τα ευρωπαϊκά μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν. Μπορούμε να δούμε στην όλη πολιτική διαδικασία την πτυχή για την που αφορά την διαβούλευση, τις αποφάσεις, ε, το, το χρόνο από, την, από τότε που λαμβάνεται η απόφαση μέχρι να εφαρμοστεί. Μπορούμε να δούμε λοιπόν χρονικά πόσο διαρκεί όλο αυτό. Ε, τα αποτελέσματα είναι αρκετά μικρά σε χρονική ε, ισχύ ε, σε σχέση με τις συνέπειες που έχουν. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ήταν καλή η χρονική διαδικασία που προτιμήθηκε. Μιλούμε για συγκεκριμένους για συγκεκριμένο κύκλο ζωής, μιλούμε για συγκεκριμένου προπολογισμού και βεβαίω διαρκέσουν όσο διαρκεί η κρίση. Θα δείτε και έναν πίνακα που δείχνει τα διάφορα έτη όπου εφαρμόστηκαν τα μέτρα αυτά, τα περισσότερα ήταν, εφαρμόστηκαν το 2009 και για τις περισσότερες χώρες τα 2010. Για την ε, εφαρμογή και για το ενέξοδο από τα μέτρα αυτά έχουμε μελετήσει την περίπτωση του Βαλγίου και της Ολλανδίας και εκεί φαίνεται ότι το phase out, η έξοδος δηλαδή, από ότι, παρόλο που βλέπετε από πριν, δεν είναι τόσο συγκεκριμένη όσο φαίνεται. Αρκετά μέτρα έχουν ε, επεκταθεί και στις δύο χώρες και το βλέπουμε αυτό και σε άλλες χώρες. Και αυτό βεβαίως ε, ε, οφείλεται και στην κρίση που ακόμη σοβεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ε, άλλοι, λόγοι, ας πούμε, οι πολιτικές επαφές ε, έχουν πάντα ρόλο να παίξουν όταν μιλούμε για τέτοια μέτρα διακριτική αφιέριας Αλλά συνολικά μπορούμε να πούμε ότι η χρονική στιγμή ήταν αρκετά καλή, αλλά το phase out ακόμη δεν έχει εφαρμόζεται μάλλον ακόμη, οπότε δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονική περίοδος για το πότε θα εφαρμοστεί. Η σύγκριση μεταξύ τώρα είπα και Ευρωπαϊκή Ένωση θα την αναλάβει ο συνάδελφος. Θα συνεχίσω με την αυτόματη σταθεροποίηση και σε σχέση με τα ε, θέματα διακριτικής ευχέρειας ως προς τα φορολογικά. Εδώ δεν υπάρχει ε, θέμα ως προς τους σταθεροποιητές, διότι όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν δύο διάβλοι. Καταρχήν υπάρχει ένας προοδευτικός χαρακτήρας στις περισσότερες χώρες και υπάρχουν και επιδόματα ανεργίας που ισχύουν αυτόματα. Άρα τι κάνουμε. Ε, βλέπουμε τα αυτόματα μέτρα και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ε, εισόδημα γενικότερα. Δηλαδή έχουμε μία μείωση του 5% που ονομάζουμε income shock και ένα 5% που αφορά το σοκ της, της ανεργίας. Ως προς τη... την μέθοδο που χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούμε την μικροπροσωμείωση που είναι το ε, μοντέλο Euromod και το Taxim. Βασιζόμαστε ε, δηλαδή σε συστήματα για να μπορέσουμε να ορίσουμε το εισόδημα. Άρα μπορούμε να φτάσουμε στην σταθεροποίηση του εισοδήματος που αντιμετωπίζουμε μετά από αυτά τα σοκ εισοδήματος και ως προς τα αποτελέσματα με βάση αυτό το ε, μαθηματικό μοντέλο βρίσκουμε ότι με ένα αναλογικό σύστημα υπάρχει σταθεροποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 32% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 38% στις ΗΠΑ. Βλέπουμε δηλαδή ε, κατά πόσο υπάρχει μία αντιστάθμιση. η, ε, αυτό το 6% είναι χαμηλό διότι βλέπουμε ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση σε σχέση με τις ΙΠΑ. Υπάρχει λοιπόν μία διαφοροποίηση. Τώρα, σε σχέση με το σοκ της ανεργίας, βλέπουμε ότι η διαφορά μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται σταθερά. Έχουμε λοιπόν μία σταθεροποίηση εισοδήματος στις τάξεις του 47% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 34% στις ΙΠΑ. Και Βεβαίως, τα επιδόματα ανεργίας διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για τη σταθεροποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ε, απορροφούν το 19% του σοκ ανεργίας σε σχέση με, ε, στην Ευρώπη σε σχέση με ένα 7% στις ΗΠΑ. Σε σχέση τώρα με την κατανομή των χώρων βλέπουμε ότι η αυτόματη σταθεροποίηση ε, διαφέρει μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Βλέπουμε λοιπόν μεγάλη ετερογένεια. Ως προς τους αυτόματους σταθεροποιητές βλέπουμε ότι είναι σχετικά ε, χαμηλή στις ανατολικές και ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο μας εκπλήσει από πλευράς ασφάλισης, διότι σημαίνει ότι τα νοικοκυριά είναι πιο ε, ευάλωτα στα σοκ εισοδήματος στις ε, ε, βόρειες χώρες βρίσκουμε μεγαλύτερη σταθεροποίηση όπως στη Δανία καθώς και χώρες της Δυτικής Ευρώπης τις επιπτώσεις στις πολιτικές μας βλέπουμε ότι τα επιδόματα ανεργίας είναι ύψης της σημασίας και ε, εξηγούν τις διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ και βλέπουμε ότι οι αυτόματοι σταθεροποιητές είναι πολύ αστάθμητοι στην Ευρώπη. Τώρα σε σχέση με την αυτόματη σταθεροποίηση είναι σίγουρα καλύτερη και εμείς ως οικονομολόγοι λέμε ότι υπάρχουν επιπτώσεις ως προς τα κίνητρα. Γι' αυτό θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτή η ανάλυση ε, δεν είναι ρυθμιστικού χαρακτήρα, αλλά είναι θετική. Ως προς τις φορολογικές επιπτώσεις, αυτό που αναλύουμε σχετίζεται με το εξής. Ορισμένες χώρες υπέστησαν φορολογικές επιβαρύνσεις κατά την χρηματοπιστωτική κρίση. Και ένα από τα αποτελέσματα είναι ότι βλέπουμε μια αρνητική σχέση μεταξύ του χρέους και του ελλείμματος που ίσχυε πριν από την οικονομική ε, κρίση και τα μέτρα τα φορολογικά που είναι μέτρα διακριτικής ευχέρειας. Αυτό δείχνει ότι οι ορισμένες χώρες υπέστησαν πίεση κατά την οικονομική κρίση καταλαβαίνουμε ότι οι φορολογικές εξισορροπήσεις και τα ε, επίπεδα χρέους επηρέασαν πολύ την κατάσταση, άρα αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να επαναληφθεί στο εγγύς μέλλον το οποίο γίνεται σαφές αν δείτε και την επόμενη διαφάνεια όπου κάνουμε προβολές για το 2015. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που κάνουν μία προβολή των ελλημάτων 5% και χρέος που φτάνει το 100% περίπου στο, του ΑΕΠ. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα άλλο ζήτημα που μας ζητήθηκε να αναλύσουμε είναι ο ρόλος των διαφορετικών επιδομάτων ανεργίας, οι διαφορετικές κοινωνικές οικονο, οικονομικοκοινωνικές ομάδες. Αρχικά κάνουμε μία σύγκριση του συστήματος πρόσβασης στα επιδόματα ανεργίας, πώς διαφορετικές εργασιακές συμβάσεις μπορούν να δώσουν ε, δικαίωμα πρόσβασης ε, σε τέτοια δικαιώματα, τι ίσχυε πριν από την κρίση και τι ίσχυε μετά την κρίση βλέπουμε ότι πολλές φορές τα συστήματα επιδομάτων ενεργείας είναι πολύ πιο κλειστά και περιοριστικά σε σχέση με τα συστήματα ελαχίστου μισθού. Και υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες ε, δεν προβλέπουν συγκεκριμένα συστήματα κοινωνικής ε, προστασίας για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν καταφέρουν να έχουν πρόσβαση στα επιδόματα ανεργίας. και έχουμε και κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπουν για αυτούς τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Στη συνέχεια προσπαθούμε να δείξουμε τις διαφορετικές ε, διαστάσεις που μπορούν να υπάρχουν ε, στην αγορά εργασίας της Ευρώπης, ποια είναι η κατανομή που υπάρχει όσον αφορά τη συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ποια είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ ε, ανεργίας και ασφαλιστικών επιδομάτων. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά που αφορούν τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα δευτερογενές τμήμα της ε, αγοράς εργασίας. Θέλουμε ουσιαστικά να δούμε εδώ πέρα ποια είναι τα προβλήματα που εντοπίζονται πολλές φορές στα συστήματα κοινωνικής υποστήριξης και στα συστήματα επιδομάτων ενεργείας. Ένα πολύ θετικό μέτρο το οποίο εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης φαίνεται στη διαφάνεια αυτή σε συνδυασμό με άλλα προσωρινά μέτρα τα οποία ελήφθησαν. Βλέπουμε όμως ότι ε, πολλές φορές τα... οι συμβάσει ορισμένου χρόνου δεν ε, εντάσσονται απαραίτητα στα συστήματα αποδοχών όσον αφορά τους ανέργους, επιδομάτων ανεργίας, τα οποία συνήθως προβλέπονται για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου. Καταλήγουμε έπειτα σε κάποιες συστάσεις όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση και τη σταθερότητα της οικονομίας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε βέβαια ότι τα μέτρα αυτά συνοδεύονται και από ένα συγκεκριμένο τίμημα, ότι πολλές φορές έχουμε κάποιες δημοσιονομικές επιπτώσεις. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία λαμβάνονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία τελικά ενισχύουν πολύ περισσότερο τους ήδη εργαζόμενους, αυτούς που βρίσκονται σε πιο ασφαλή συμβάση εργασίας, ενώ αντίθετα πιο εκτεθειμένοι είναι τελικά οι αυτοαπασχολούμενοι, οι άνθρωποι που εργάζονται στα πλαίσια μια σύμβαση ορισμένου χρόνου. Βλέπουμε επίσης ποια θα ήταν τα θετικά ωφέλη ενός συστήματος αυτοματοποιημένης ε, σταθεροποίησης και πώς μπορούμε να μειώσουμε τη διακριτική μεταχείριση κατά των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχει απασχολήσει συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Ένα άλλο πόρισμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι είναι θετική βέβαια η αυτόματη σταθεροποίηση, αλλά εμπεριέχει και κάποιο τίμημα είναι σημαντικό να λάβουμε δηλαδή υπόψη μας τις δημοσιονομικές επιπτώσεις ενός τέτοιου συστήματος. Το ίδιο ισχύει και για τα μέτρα αυτά τα οποία μπορούν να λάβουν, ε, ε, τα οποία εξαρτώνται από διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων, που μπορούν να αποφέρουν πολύ θετικά αποτελέσματα γρήγορα, αλλά έχουν και αυτά συγκεκριμένε δημοσιονομικέ αρνητικέ επιπτώσει. Πολλές φορές τα μέτρα αυτά συνδέονται με συγκεκριμένους δείκτες όπως η αύξηση της απασχολησιμότητας για παράδειγμα. Τα μέτρα αυτά επίσης έχουν ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και πολλές φορές μετά από την πάροδο συγκεκριμένων ετών βαθμιαία καταργούνται. Όσον αφορά το κοινοτικό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρούμε ότι εδώ πέρα μπορεί να διαδραματιστεί ένα συγκεκριμένο ρόλο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μπορούσε να ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν συντονισμένα συστήματα κοινωνική προστασία. Θα μπορούσε επίση να επέμβει θετικά στι αγορέ εργασία των κρατών μελών. Είναι πολύ σημαντικό επίση να υπάρχει ένα σύστημα αυτόματης σταθεροποίησης που θα επιτρέπει σε όλα τα κράτη-μέλη συντονισμένα να αντιδρούν κάθε φορά που ε, προκύπτει μια οικονομική κρίση. Επίσης είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση συντονισμένα να αξιολογούμε την εξέλιξη της αγοράς εργασίας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου και η ανταπόκριση έπειτα να είναι πολύ πιο συντονισμένη και κοινή και να μην είναι κατακαιρματισμένη απομονωμένη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε για την πλήρη αυτή παρουσίαση. Μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. κυρία Μωρά έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, είπατε ότι ήταν ιδιαίτερα πλήρης η παρουσίαση αυτή. Πρέπει να σας πω ότι είμαι κάπως απογοητευμένη. Καταρχάς, σκέφτομαι τους διερμηνείς, οι οποίοι χρειάστηκε να παρακολουθήσουν μια παρουσίαση πάρα πολύ γρήγορη και πυκνή, μεστή. Δεν ήταν λοιπόν εύκολη η δουλειά τους. Βλέπω όμως το τέτοιο κείμενο το οποίο μας έχει δοθεί και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη όταν βλέπω ότι η μελέτη αυτή βασίζεται σε γραφικές παραστάσεις οι οποίες είναι εντελώς δυσνόητες, δεν μπορούμε καν να τις διαβάσουμε με τον τρόπο που είναι τυπωμένες. Σίγουρα, αν είχαμε εδώ πέρα λίγο χρώμα, θα καταφέρναμε να τι καταλάβουμε καλύτερα. Αλλά έτσι όπω είναι τυπωμένε, ασπρόμαυρε, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από τι γραφικέ αυτέ παραστάσει. κατέβαλα φοβερέ προσπάθειε για να τι καταλάβω, αλλά ό,τι και να έκανα δεν κατάφερα να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα διαβάζοντα αυτέ τι γραφικέ παραστάσει. Δεν μπορώ καν να δω τις γραμμές ξεκάθαρα, δεν μπορώ να δω τις καμπύλες, δεν, δεν καταλαβαίνω ποια καμπύλη αντιστοιχεί σε ποια χώρα. Σας λέω λοιπόν για άλλη μια φορά ότι είμαι ιδιαίτερα απογοητευμένη και εκφράζομαι με τον τρόπο αυτό γιατί ε, ουσιαστικά το κείμενο αυτό δεν βοηθά καθόλου τους συντάκτες της ε, μελέτης αυτής, το την παρουσίαση προσπάθησα να κάνω. Ε, ε, συγγνώμη, θα ήθελα να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, λέει η ομιλήτρια προσπαθούσα να δω πού προβαλόταν η παρουσίαση αυτή. Δεν κατάφερα να δω τίποτα γιατί περίμενα να δω τουλάχιστον τι γραφικές παραστάσεις σε διαφάνειες έγχρωμες. Ενδεχομένως οι συναδελφοί μου να είναι πιο ικανοί από μένα και να κατάφερα να καταλάβω. Εγώ πάντως δεν το κατάφερα. Βασίστηκα στο κείμενο αυτό τέλο πάντων, καθώ επίση και στι συστάσει χάραξη πολιτική που γίνονται στο τέλο. Και ειλικρινά τι να σας πω, τα όσα λέγονται εδώ πέρα, όσον αφορά την σταθεροποίηση, όσον αφορά την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους προσωρινά απασχολούμενους και τους μόνιμους εργαζόμενους, πραγματικά δεν κατάφερα να δω κάτι το ιδιαίτερα επαναστατικό εδώ πέρα, δηλαδή τίποτα διαφορετικό σε σχέση με τις μελέτες που έχουμε εξετάσει στο παρελθόν. Η μελέτη αυτή δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει σε μία μελλοντική επικοδομητική συζήτηση που θα έπρεπε να λάβει χώρα. Στις, στα συμπεράσματα βλέπουμε ότι η κρίση συνέβαλε στην επιτάχυνση της αλλαγής των κοινωνικών συστημάτων στα κράτη-μέλη. Ναι, αυτό το είδαμε όλοι. Ωστόσο, τίθεται ένα ερώτημα το οποίο θα έπρεπε να υποβάλλουμε στους συντάκτες της μελέτης. Δεν θα έπρεπε κάπου εδώ πέρα να λέγεται ότι πρέπει να αυξηθεί η κοινωνική προστασία στα κράτη-μέλη αλλά να μειωθούν οι κερνητικές επιπτώσεις στον προπολογισμό. Συμφωνώ αν θέλετε με τη σύσταση αυτή, αλλά πώς μπορούμε να μειώσουμε το επίπεδο κοινωνικής προστασίας σε χώρες που παραδοσιακά έχουν ένα πολύ δυνατό σύστημα κοινωνικής προστασίας, σε χώρες που παραδοσιακά λειτουργούν με τον τρόπο αυτό. Παρ' αυτά απάντηση στο ερώτημά μου αυτό δεν κατάφερα να δω. Ήθελα απλώς ε, να σας πω ότι οι συγγραφείς της ε, μελέτης δεν είναι υπεύθυνη για το γεγονό ότι έχει τυπωθεί το έντυπο ε, σε, έχει, είναι μαυρό άσπρο τέλος πάντων και όχι έγχρωμο. Οι υπεύθυνοι είναι οι κοσμήτορες. Oui, mais vous, aurez évidemment par courriel euh, la version euh, couleur. Ε, δυστυχώς το τυπογραφείο δεν μπορούσε να τυπώσει μία έγχρωμη έκδοση. Εν πάση περιπτώσει δεν φέρουμε εμείς την ευθύνη. Θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο. Bien. Ε, χωρίς μικρόφωνο μιλητής, δεν τον ακούμε. Uh, sorry, I saw the green... Α, με συγχωρείτε. Um, just it arises from, from, from a... uh, η κυρία Όκνη είπε για τις, μίλησε για τις δυσκολίες του να μετακινηθούν οι άνθρωποι από την ευημερία, από την, το, μια πολιτική ευημερία στην απασχόληση εκ νέου. Θα θέλαμε ένα σύστημα πρόνοιας να μειώσει τις παγίδες φτώχειας. Πολλά συστήματα βασίζονται στο εισόδημα, στην εισοδηματική πολιτική. Δηλαδή οι άνθρωποι επειδή έχουν χαμηλόμισθες, εργασία χάνουν πολλά. Άρα δεν θέλει κανείς να μετακινηθεί σε ένα τέτοιο σχήμα και να χάσει τα οικογενειακά πλεονεκτήματα. Άρα θα πρέπει να ξεφύγουμε από τις παγίδες φτώχειας και να προωθήσουμε αξιοπρεπή εργασία. Και νομίζω ότι αυτό αφορά ένα συντονισμό, γενικότερο συντονισμό γιατί δεν μπορούμε να ε, προβάλλουμε ένα αυτοκαταστροφικό σύστημα όταν μιλάμε για κοινωνική απασχόληση έναντι της εργασίας. Ξέρω ότι υποστηρίζετε αυτή την ιδέα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τονιστεί υπό την έννοια αυτή της συζήτησης. Η κυρία Φιγκεϊρέτο. Ευχαριστώ. Λυπάμαι γιατί δεν μπόρεσα να παρευρεθώ νωρίτερα, αλλά συμμετείχα στη μεγάλη διαδήλωση που λαμβάνει η χώρα έξω από το κτίριο αυτό και διαμαρτυρηθήκαμε γιατί δυστυχώς έρονται πολλά πλεονεκτήματα στους εργαζόμενους. Στη χώρα μας είχαμε ένα επίδομα ανεργίας που κάλυπτε κάπως τους ανέργους αυτή τη στιγμή ε, εξαιτίας αυτής της νέας πολιτικής μειώθηκε ο χρόνος χορήγησης του επιδόματος ανεργίας και πάνω από 40% των ανέργων δεν έχουν καμία αποδοχή, δηλαδή κανένα επίδομα. Επίσης, το κοινωνικό επίδομα επανεισδοχής στο χώρο εργασίας είναι 189 ευρώ το άτομο, δηλαδή είναι γελίο. Ε, θα ήθελα μερικοί από εμά να προσπαθήσουν να επιζήσουν ένα μήνα με 189 ευρώ για να πληρώσουν τα πάντα, δηλαδή στέγη, τροφή, ιατρικά έξοδα, μεταφορές, εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Αυτό τι σημαίνει έμπρακτα. Σημαίνει ότι ο δείκτης φτώχειας αυξάνεται δραματικά. Άρα πού βρίσκεται η κοινωνική Ευρώπη, πού βρίσκεται η κοινωνική και η οικονομική συνοχή, πώς είναι δυνατόν να επιβάλλουμε μέτρα, μέτρα τόσο αυστηρά με βάση το σύμφωνο σταθερότητας χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι η χώρα μου. Και έτσι να πολλαπλασιάζεται η φτώχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πού καταπολεμούμε τη φτώχεια. Αυτό το ερώτημα θα ήθελα να θέσω. Γιατί χρειαζόμαστε ε, απασχόληση. Εάν όμως ε, δεν υπάρχει, πώς θα αφήσουμε τους ανθρώπους, σε τι κατάσταση. βρίσκονται σε κατάσταση ε, επαυξημένης φτώχειας και δραματικής φτώχειας. Μιλάμε για ελάχιστο μισθό που βρίσκεται στο κατόφλι της φτώχειας κατά την άποψή μου. Θα ήθελα να ξέρω τι πιστεύουν οι εμπειρογνώμονές μας. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Φαίνεται πως όχι. Θα ήθελα οι προσκεκλημένοι μας να απαντήσουν. Euh, Δεν ξέρω ποιος θέλει το λόγο από τους τρεις. Να ξεκινήσω εγώ και να δούμε μετά αν μπορούν να με στηρίξουν και οι συνάδελφοι. Καταρχήν νομίζω ότι έχει γίνει κάποια παρεξήγηση. Όχι μόνο για την εκτύπωση των διαφανειών, αλλά και για την κοινωνική προστασία. Προφανώ εμεί δεν είμαστε ενάντια στην κοινωνική προστασία. Δεν είπαμε ποτέ τέτοιο πράγμα. Αλλά ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνάς μας είναι ότι η κοινωνική προστασία δεν είναι μόνο ενδιαφέρουσα ως στόχος κοινωνικής πολιτικής, αλλά ως και ως στόχος οικονομικής πολιτικής, γιατί προσπαθεί να συνδυάσει και την αγορά εργασίας και την οικονομία και να καταλήξει σε κάποια, σε κάποια ωφέλεια κατά τη διάρκεια της κρίσης. Μιλούμε για πρόσβαση σε διάφορα επιδόματα κοινωνική ενίσχυση. Ε, αυτό όμω επαφείται στα κράτη-μέλη και στην νομοθεσία του. Οπότε γι' αυτό μιλούμε για, την, για τον καθαρισμό κάποιων προγραμμάτων ε, ελάχιστων επιδομάτων, ε, επιδότηση δηλαδή με ελάχιστα επιδόματα είτε ανεργία είτε οτιδήποτε άλλο είναι αυτό. Ή ασφάλεια κατά τη διάρκεια τη ανεργία Ιδιαίτερα όταν μιλούμε για άτομα ε, μικρής ηλικία ή γυναίκες που ξεκινούν τη δουλειά και που πρέπει να έχουν κάποια ενίσχυση, κάποια επιδότηση. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τα περισσότερα κράτη-μέλη που πρέπει να ε, ξαναπροσδιορίσουν την κοινωνική πολιτική τους έτσι ώστε να έχουμε ένα εργαλείο που να μας ε, βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε δυσκολίες προκύψουν στο μέλλον. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο αυτό. Συμφωνώ βεβαίως απόλυτα και ε, με αυτά που είπε η κυρία Φιγκερέιδο από την Πορτογαλία. Προφανώς πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα ενίσχυσης ώστε να προστατεύονται οι πολίτες ενάντια στην... να προστατεύονται οι πολίτες από τη φτώχεια. Τα κοινωνικά προγράμματα θα πρέπει να συνδυάζονται και με ε, ε, σωστές λειτουργικές πολιτικές για την αγορά εργασίας. Συμπεριλαμβάνοντας βέβαια και προγράμματα κατάρτισης ίσως και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό δεδομένου ότι οι, αυτές οι περίεργες ε, καταστάσεις που ζούμε συνήθως αλλάζουν δραματικά την οικονομική κατάσταση μιας χώρας και το ίδιο ισχύει και για την αποφυγή ε, των, ε, της φτώχειας μέσω κινήτρων. Η εργασία επιπληρωμή θα πρέπει να είναι πολύ πιο ελκυστική πάντα από οποιοδήποτε επίδομα ανεργίας ώστε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο του να βρεθούν ε, σε ε, κατάσταση φτώχειας ε, και άλλοι, και άλλοι πολίτες στο μέλλον. Αν υπάρχουν άλλα σχόλια, ευχαριστώ να απαντήσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω για την κατάσταση της Πορτογαλίας διότι από ό,τι κατανόησα ε, βλέπω ότι δεν γνωρίζετε τι συμβαίνει στην Πορτογαλία, ποια είναι τα κοινωνικά μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης σε σχέση με ένα ελάχιστο εισόδημα ε, για όλες τις φτωχές οικογένειες υπάρχει και επίδομα ανεργίας μακράς διαρκείας, καθώς και συμπληρωματικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν πρόσφατα. Είναι σαφές ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού και με το σύμφωνο σταθεροποίησης επιβάλλεται στις κυβερνήσεις να μειώσουν αυτή την κοινωνική στήριξη. Δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζετε την κατάσταση πραγματικά όπως ισχύει στην Πορτογαλία. Σας ευχαριστώ. Euh, θα ήθελα οι εμπειρογνώμονες να μου πούν κατά πόσο ξέρουν την κατάσταση στην Πορτογαλία, δεν την ξέρουν και μετά θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Um, screened um, all that... Ξέρουμε ότι έχουν ληφθεί κάποια εθνικά μέτρα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεμονωμένα. Ξέρουμε επίσης ποιο είναι το πρόγραμμα στην Πορτογαλία, αλλά ξέρουμε π.χ. ότι είναι τελείως διαφορετικό το πρόγραμμα αυτό από ό,τι σε άλλες χώρες, όπως η Ιταλία. Γνωρίζουμε την περίπτωση της Πορτογαλίας, αλλά εσείς το την ξέρετε καλύτερα από εμάς. Νομίζω ότι θα κλείσουμε αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης εδώ. Θα σας αποστείλουμε τη μελέτη σε, ε, μέχρι το τέλος του μήνα, λέει η Πρόεδρος σε λίγο χρονικό διάστημα, όταν δοθεί η τελική μορφή και θα διακόψουμε τις εργασίες μας για να περάσουμε απέναντι και θα βρεθούμε εδώ αύριο το πρωί στις 9. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.